βάση της ημερήσιας διάταξης προχωρούμε στην δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την προετοιμασία της Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης Κορυφής. Θα δεις, δώσω αμέσως το λόγο στην κυρία Χένης Πλασάρτ εξ ονόματος του Συμβουλίου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξεκινώ λέγοντας ότι κατά άποψή μου η Σύνοδος Κορυφής είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει η παγκόσμια κοινότητα να χάσει την Πέμπτη τα συμπεράσματα, αναμένονται να υιοθετηθούν τα συμπεράσματα από το συμβου, για το Συμβούλιο, για την Σύνοδο Κορυφής από το Συμβούλιο, ενώ προετοιμάζεται και μια κοινή θέση της Ένωσης και των κρατών σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Το... Η Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφής θέλουμε να είναι επιτυχία. Ήδη από τον Ιούλιο έχουμε ξεκινήσει με έναν απεσταλμένο για, το, για την ε, διάσκεψη κορυφής, ούτως ώστε να έχουμε μόνιμη επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, διεθνείς οργανισμούς, ΟΗΕ, κράτη-μέλη, άλλα κράτη-μέλη και άλλους φορείς. Θέλω να αναφερθώ σε κάποια από τα σημαντικότερα θέματα που θέλουν να προκύψουν από τη διάσκεψη κορυφής τα κράτη-μέλη. Θέλουμε η παγκόσμια κοινότητα να δεσμευτεί εκ νέου στις αρχές ε, της ε, του ανθρωπισμού, της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας. Επίσης, να αντιμετωπίσουμε τις βασικές ε, αιτίε της ανθρωπιστικής κρίσης, επιλύοντας με ειρηνικό τρόπο τις σειράξεις, προλαμβάνοντας την γένεση των συγκρούσεων. Θέλουμε όλες οι πλευρές να σέβονται, σε ε, μια σύγκρουση να σέβονται το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Και θέλω να επαναλάβω αυτό που είπα κατά τη συζήτησή μας ε, στις Βρυξέλλες πριν από δύο εβδομάδες. Η επίθεση σε δομές όπως νοσοκομεία και σχολεία είναι απαράδεκτη θα πρέπει η ανθρωπιστική νομοθεσία, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο να είναι ψηλά στην ημερήσια διάταξή μας και να μιλούμε σαφώς κατά σοβαρών παραβιάσεων. Η τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου συνδέεται επίσης και με ένα βασικό θέμα της Συνόδου Κορυφής. Να βάλουμε τον άνθρωπο στο κέντρο της ανθρωπιστικής δράσης. Πρέπει να απομακρυνθούμε λοιπόν από την, ε, τα γραφεία σχεδιασμών στις πρωτεύουσε και να ακούμε τους πληθυσμού που πλήττονται. Ταυτόχρονα να προχωρήσουμε στην ε, εκρίζωση της ε, βίας που, που σχετίζεται με το φύλλο και να μην ε, αντιμετωπίζουμε τις γυναίκες μόνο ως θύματα αλλά ως και άμεσα βασικούς εμπλεκόμενους φορείς σε όλες τις ανθρωπιστικές αντιμετωπίσεις. Η Προεδρία πιστεύει επίσης ότι μπορούμε να πετύχουμε καλύτερη ανθρωπιστική παρέμβαση προωθώντας την καινοτομία στην χρηματοδότηση ε, των ανθρωπιστικών δράσεων, των νέων τεχνολογιών, των νέων εταιρικών σχέσεων. Σαν παράδειγμα της τελευταίας ε, πρότασης, η Ολλανδία μετέχει στην Παγκόσμια Συμμαχία για την Ανθρωπιστική Καινοτομία που θα ξεκινήσει στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο της διάσκεψης κορυφής. Να πω επίσης και δύο λόγια για την ανθρωπιστική χρηματοδότηση. Η Ολλανδία και άλλα κράτη-μέλη βρίσκονται μεταξύ των 15 μεγαλύτερων δωρητών σε παγκόσμιο επίπεδο. Μαζί με την Τουρκία οι δωρητές κλήθηκαν στο High Level Panel ανθρωπιστικής χρηματοδιώτησης για να διαπραγματευθούν την αποτελεσματικότητα των δυνατοτήτων χρηματοδότησης με τις μεγαλύτερες οργανώσει υλοποίηση. Εμεί είχαμε την πρώτη τέτοια συνάντηση στι 29 Φεβρουαρίου στο Άμστερνταμ. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, μαζί με την Παγκόσμια Τράπεζα, ξεκινήσαμε τη συζήτηση για τη διαφάνεια των ενισχύσεων. Και θέλω να ευχαριστήσω εκ νέου την Επιτροπή και το Ηνωμένο Βασίλειο που φιλοξένησαν τη δεύτερη συνάντηση των Σέρπαν. Η τελευταία τέτοια συνάντηση με τη Σουηδία συνεχίζεται αυτή τη στιγμή στην Νέα Υόρκη, μπορεί να το ξέρετε. Ελπίζουμε να υπάρχει μια γρήγορη ε, έκβαση. Ως Προεδρία του Συμβουλίου θέλουμε όσο περισσότεροι δωρητές και ανθρωπιστικές οργανώσεις να μετάσχουν σε αυτή τη συνολική συμφωνία και τις ε, δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται. Θέλω να ευχαριστήσω κλείνοντα το Κοινοβούλιο για το ενδιαφέρον που έχει δείξει, τις συμβουλές που παρέσχε. Η συμμετοχή σας είναι σαφής απόδειξη των δεσμεύσεων και της αφοσίωσής σας και περιμένω να ακούσω περισσότερα πράγματα από αυτά που εσείς προσδοκάτε από την διάσκεψη ορυφής εν ώψη της Φιωτινούπολης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το, το λόγο τώρα έχει ο κ. Κυλιανίδης. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, κυρία Υπουργέ, Μόνο 12 μέρες μας ε, χωρίζουν από την ε, διάσκεψη κορυφής. Είναι μια ευκαιρία ολόκληρης γενιάς να κάνει τη διαφορά, να κάνει την ιστορία, να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλο τον κόσμο ότι η παγκόσμια ανθρωπιστική βοήθεια χρειάζεται δράση, συλλογική δράση. Η διάσκεψη κορυφής δεν μπορούσε να είναι πιο επίκαιρη. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε είναι τεράστιες. Πέρσι βοηθήθηκαν με ανθρωπιστική βοήθεια πάνω από 100 εκατομμύρια άνθρωποι. Είναι οι, μετα, μετακινήσεις πληθυσμών οι μεγαλύτερες μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Εκατομμύρια εγκαταλείπουν τις εσκηριστίες τους για να αποφύγουν τις καταστροφές από την κλιματική αλλαγή και οι άνθρωποι φεύγουν για πολύ μεγαλύτερα διαστήματα από ό,τι ποτέ στο παρελθόν. Ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρινόμαστε στις αυξανόμενες ανάγκες δεν είναι πλέον ε, ε, βιώσιμος. Οι άνθρωποι που ε, πλήττονται από τις κρίσεις πρέπει να φύγουν με αξιοπρέπεια και όχι απλώς να δέχονται βοήθεια. Δεν μπορεί να συνεχίσουν τα πράγματα ως έχουν. Η ασχολούμενοι με την ανθρωπιστική βοήθεια εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες και συνεχίζουν παρά τη δράση τους. Όμως θα πρέπει να εμπλακούν και άλλοι παράγοντες ώστε το ανθρωπιστικό σύστημα να είναι πιο αποδοτικό, πιο αποτελεσματικό αλλά και για να προληφθούν οι συγκρούσεις, να μειωθεί ο κίνδυνος καταστροφών και να αυτονομηθούν κοινότητες. Δεν είναι μυστικό ότι είχαμε μεγαλύτερες προσδοκίες για και καλύτερα πολιτικά αποτελέσματα, για καλύτερα πολιτικά αποτελέσματα από αυτή τη διάσκεψη κορυφής. Παρά τα αυτά, ελπίζω ότι τελικά θα μπορέσουμε να δώσουμε ένα ωραίο, ένα ισχυρό όραμα μετά τη διάσκεψη κορυφής. Ε, η δράση αυτή είναι πολύ καλή βάση για περαιτέρω κινητοποίηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει να συνεχίσει να παίζει το ρόλο της σύμφωνα με αυτά τα οποία διατυπώθηκαν στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής μάλλον το ψήφισμα για την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής που ενέκρινε το Δεκέμβριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναγνωρίζουμε τη δική σας συνεισφορά στη διατύπωση των προτεραιοτήτων μας και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα που τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συμμετέχουν στην διάσκεψη κορυφής. Η συμμετοχή σας είναι σημαντική για μας και συνεννοηθήκαμε τα Ηνωμένα Έθνη στο ανώτατο επίπεδο για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή σας. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση πηγαίνουμε στη διάσκεψη κορφής με τρεις ξεκάθαρους τόκους. και θα ήθελα να ευχαριστήσω την παρούσα Προεδρία αλλά και τις προηγούμενες και άλλες Προεδρίες γι' αυτό. Πρώτον, έλλειψη σεβασμού του διεθνούς ανθρωπιστικού, στο ανθρωπιστικό δίκαιο αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο. Οι πολίτες γίνονται στόχος, καταστρέφονται ιατρικές εγκαταστάσεις και σχολεία και τα όσοι ασχολούνται με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας πλήττονται. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Θέλουμε λοιπόν να στηριχθούν οι αξίες και οι αρχές ε, της ανθρωπιστικής βοήθειας. Είμαστε υπέρμαχοι του ε, σεβασμού του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και θέλουμε η διάσκεψη κορυφής να επαναλάβει τη σημασία του. Χαιρετίζω ιδιαίτερα το πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για σχετικά με τις ε, επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία γιατί επαναλαμβάνει αυτή την προτεραιότητα του ανθρωπιστικού δικαίου. Δεύτερον, να εξασφαλίσουμε πιο αποτελεσματική ανθρωπιστική δράση. Ο ανταγωνισμός πρέπει να αντικατασταθεί από την συνεργασία ανάμεσα στους ε, ε, οργανισμούς οι οποίοι εργάζονται για αυτό το σκοπό. Και βεβαίως πρέπει να εμπλέκονται να εμπλέκεται και ο ιδιωτικό τομέα. Για το σκοπό αυτό έχουμε ξεκινήσει συζητήσεις για τη συνέχιση της, ε, της δράσης έκθεσης του ε, υψηλού επίπεδου ανθρωπιστικής βοήθειας. Τέλος, θέλουμε να ενισχύσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια και να εμπλακούμε πιο ε, δυναμικά με τους ε, εταίρους μας. Καταστάσεις παρατεταμένης απομάκρυνσης από τις αιστείες συνεπάγεται ότι οι άνθρωποι πρέπει από εξαρτώμενοι από τη βοήθεια να μπορέσουν να γίνουν αυτόνομοι. Αυτό είναι ο τελικός στόχος ε, της βασικής δέσμευσής μας. Η ανακοίνωσή μας για την βίαιη μετακίνηση που εγκρίθηκε στις 26 Απριλίου θα ασχοληθεί θα ασχοληθούμε με αυτά τα βασικά ζητήματα και σκοπεύουμε να καταλήξουμε σε σοβαρές δεσμεύσεις. Περιμένουμε και από τους άλλους να κάνουν το ίδιο. Για την επιτυχία της διάσκεψης κορφής πρέπει να αναλυφθούν πολιτικές δεσμεύσεις στο ανώτατο δυνατό επίπεδο, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την αποτελεσματική συνέχιση τις προσπάθειες. Η διάσκεψη κορυφής δεν θα αποτελέσει μόνο το, την αποκορύφωση προετοιμασίας και συζητήσεων που διήρκεσαν μήνες ολόκληρους. Θα είναι και το ξεκίνημα της ε, αλλαγής του διεθνούς ανθρωπιστικού συστήματος κυρίως μέσω της υλοποίησης των δεσμεύσεων που θα αναλάβουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσουμε τους, με τους ομιλητές από τις πολιτικές ομάδες. κυρία Ζαμπόρσκα είναι η πρώτη, η οποία δεν είναι παρόν βέβαια, παρούσα. Ο κύριος Γκερέρος Σαλώμα από τους Σοσιαλιστές για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω καταρχήν ότι αυτή η διάσκεψη κορυφής έρχεται σε μια χρονική στιγμή μεγάλων οργανωτικών δυσκολιών. Είναι δύσκολη η παρουσία εκπροσώπων από το Ευρωπαϊκό μας Κοινοβούλιο για να είναι παρόντες στο κατάλληλο επίπεδο στη διάσκεψη κορυφής Κωνσταντινούπολης, αλλά όπως είπε και ο κύριος Επίτροπος, έρχεται σε μια απαραίτητη χρονική στιγμή, μια στιγμή απαραίτητη δράση, στην κατάλληλη στιγμή. Αυτή τη στιγμή έχει συσσωρευτεί ένα μεγάλο αριθμό κρίσεων πολύ ψηλού επίπεδου στον κόσμο από το Ιράκο στη Συρία ω το Νότιο Σουδάν, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία αλλά και στην Ουκρανία, στην Ιεμένη, στην Λιβύη και σε άλλα τμήματα του κόσμου. Αυτή τη στιγμή έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που είναι εκτοπισμένοι από τις εστίες τους περίπου 120 εκατομμύρια σε 37 διαφορετικές χώρες. Το ίμιση αυτών σχεδόν είναι παιδιά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η μεγαλύτερη απόκληση έναντι της ανάγκης να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων και της χρηματοδότησης που είναι ε, διαθέσιμη. Έχουμε μία μείωση κατά 40% της ε, χρηματοδότησης αυτής, ενώ συγχρόνως λαμβάνουν χώρα όλο και περισσότερο παραβιάσεις των αρχών της ανθρωπιστικής δράσης, επιθέσεις σε εγκαταστάσεις και σε ανθρώπους που ασκούν την ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι η κατάλληλη στιγμή λοιπόν για να κάνουμε μια σημαντική έκκληση, να δώσουμε μια σημαντική όθηση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ανθρωπιστικές κρίσεις σε όλο τον κόσμο. Υπήρξε μια σημαντική συνένεση τους ε, παγκοσμίου επίπεδου διάλογους, σε περιφερειακού επίπεδου διάλογους και πιστεύω ότι η θέση που εξέφρασε ο κύριος Επίτροπος και οι εκπρόσωπος του Συμβουλίου αντανακλούν αυτή τη συνένεση σε σχέση με το πρακτέο. Παρόλα αυτά υπάρχει λιγότερη αποφασιστικότητα σε σχέση με τις δεσμεύσεις που πρέπει να αναλυθούν. Η Κομισιόν παρουσίασε τις προτάσεις της και τις προτεραιότητές της. Το Κοινοβούλιο την υποστήριξε. Το Κοινοβούλιο επίσης ε, συνέταξε μια έκθεση όπου ζητήσαμε να υπάρξει μια συνολική συνένεση για την ανθρωπιστική δράση και όπου ζητούσαμε να υπάρξει μια καλύτερη προστασία μέσα στις πολιτικές ε, συνεργασίες για την ανάπτυξη, να προστατεύσουν περισσότερο τους ανθρώπους που είναι εκτοπισμένοι. Χρειαζόταν να υπάρχει και περισσότερος ρόλος για τους τοπικούς πληθυσμούς, για τις γυναίκες και για τους εκτοπισμένους, όπως ανέφερε η κυρία ε, υπουργό και θέλαμε να έχουμε την κατάλληλη χρηματοδότηση. Αυτό το οποίο ζητώ τώρα στην, από την Επιτροπή και το Συμβούλιο είναι η Κωνσταντινούπολη να είναι μόνο το πρώτο βήμα και να ακολουθήσουν σοβαρέ δεσμεύσει και τη Κομισιόν και των κρατών μελών ώστε να υπάρξει αυτή η συνολική συνένεση για την ανθρωπιστική δράση, για να υπάρξει μια νέα πρωτοβουλία που θέτει από κοινού την πολιτική ανάπτυξη και την ανθρωπιστική πολιτική και που να οδηγήσει σε δεσμεύσεις για την καταγγελία των παραδιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων και τις επιθέσεις στους ανθρωπιστικούς φορείς. Κλείνω κυρία Πρόεδρε λέγοντας ότι η Κωνσταντινούπολη θα πρέπει να είναι το πρώτο βήμα για να επανέλθει η αξιοπρέπεια στο απαραίτητο όριο στις ανθρωπιστικές ε, παρεμβάσεις. Ευχαριστώ κύριε λεπτό. Πόλεμοι φυσικές καταστροφές, επιστημιστική ανασφάλεια, κάποιες από τις μάστιγες του κόσμου, παντού ο κόσμος ζητά βοήθεια στη Συρία, την Ιεμένη, την Ουκρανία και την Τουρκία που ηρωνικά θα έλεγε κανείς υποδέχεται την παγκόσμια ανθρωπιστική διάσκεψη κορυφής. Ματώνει η χώρα από τη συμπεριφορά του Ερντογάν. Ζητώ από τα κράτη-μέλη να υποστηρίξουν ε, τη, τους Κούρδους και τους Τούρκους. Συμφωνούμε όλοι νομίζω ότι στην παρούσα κατάσταση η κρίση απαιτεί περισσότερα χρήματα αλλά και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Πρέπει να διδαχθούμε από τα λάθη του παρελθόντος. Ο συντονισμός είναι αναγκαίος. Η προστιθέμενη αξία των ΜΚΟ είναι σημαντική. Η ανθρωπιστική βοήθεια και η αναπτυξιακή βοήθεια πρέπει επίσης να συνδυαστούν καλύτερα. Χρειάζονται ταυτόχρονα μέτρα προληπτικού χαρακτήρα, προλαμβάνοντας δηλαδή ε, κρίσεις. Η εκ των υστέρων αντιμετώπιση των κρίσεων κοστίζει περισσότερο. Ταυτόχρονα πρέπει να μην συνδέουμε πολιτική και ασφάλεια με την ανάπτυξη θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα από τη Σύνοδο Κορυφής και συμφωνώ με τον προηγούμενο μιλητή, δεν πρέπει του χρόνου να ξαναβρεθούμε χωρίς να έχουν υπάρξει ουσιαστικές επιτόπου αλλαγές. Χωρίς αλλαγές η, σύνοδο, η διάσκεψη κορυφής θα αποτύχει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή οι οποίοι παρακολουθούν αυτές, αυτή τη διάσκεψη κορυφή καμιά φορά αισθάνε ε, ε, χαίρεται για ορισμένα πράγματα παρά το ότι υπάρχουν και πιστεύουν ότι οι καταστροφές μπορούσαν να είχαν αποφευθεί χάρη στην ε, ανθρωπιστική δράση. Υπάρχουν όμως φοβερά γεγονότα τα οποία θα θέσουν σε αμφισβήτηση τη διάσκεψη κορυφή. Πρώτον, η όλο και μεγαλύτερη απειλή κατά τη ασφάλειας των ιατρικών αποστολών. Η κρίση θεωρείται μοιραία. Και τρίτον, η δέσμευση των κρατών, κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέχει από το οικονομικό αποτέλεσμα χρηματοδότησης. Όλο και περισσότερο απειλούνται οι ε, ιατρικές αποστολές. Οφείλεται αυτό σε ανθρώπινα λάθη ή σε άλλους λόγους. τα κράτη που, που θα πάνε στην Κωνσταντινούπολη θα πρέπει να σταματήσουν την ε, αντικειμενικότητα όσον αφορά την ε, στρατιωτική επέμβαση, αυτή δεν είναι η συνήθις απάντηση. Πρέπει λοιπόν εγκαίρως να κινητοποιείται η διπλωματία. Όχι οποιαδήποτε διπλωματία, αλλά καλύτερη δυνατή. Τα κράτη που θα πάνε στην Κωνσταντινούπολη θα πρέπει να το λάβουν αυτό υπόψη τους. Οι δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι γενναιόδορες. Ε, βεβαίως ανανεώνονται συχνά, για τον απλούστο το λόγο ότι δεν έχουν τηρηθεί για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι θέμα αξιοπιστίας. Τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να το θυμούνται αυτό. Δεν αρκεί να διαπιστώνει κανείς ότι οι άλλοι, σχεδόν όλοι οι άλλοι δεν τα πάνε όσο καλά όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της. Αυτό δεν θα πρέπει να κάνει τους 28 να μειώσουν την προσφορά τους. Οι ελπίδες μας βρίσκονται στη δέσμευση της Προεδρίας και του ε, Επιτρόπου. Καλή τύχη Χρήστο. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Όρμπαν Κρέσπο για την ΚΟΕ. Ε, Κυρίες και κύριοι, δυστυχώς όλο και συχνότερες είναι οι αυτοθοπιστικές κρίσεις και η αιτία δεν είναι μόνο η αλλαγή του κλίματος ή φυσικές καταστροφές. Συχνά ένοπλες συγκρούσεις καρπή οικονομικών συμφερόντων. Επίσης, συνέπεια πολιτικών ε, αποφάσεων όπως το κλείσιμο των συνόρων μετά από την άφηξη χιλιάδων προσφύγων που οδήγησε σε ανθρωπιστική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις λοιπόν ως προς την πραγματική δυνατότητα ε, διεξόδου που θα παράσχει η σύνοδος αυτή κορυφή. Τι, ε, χρειάζονται, τι χρειάζονται οι, οι διασκέψεις κορυφής αν οι ίδιες οι πολιτικές δημιουργούν κρίσεις. Ίσως απλώς η σύνοδος, η σύνοδος αυτή να έχει στόχο να κρύψει τις ε, πολιτικές της Ένωσης, ιδίως δε του νέου εταίρου μας της Τουρκίας. Δεν χρειάζεται να δίνουμε με τα αριστερά και να δίνουμε, ε, να δίνουμε δώρα με το αριστερό χέρι και χαστούκια με το δεξί χέρι. Αν θέλετε να προσφέρετε λύσεις μπορείτε να το κάνετε αύριο. Ανοίξτε ασφαλείς δρόμους παρέχοντας έναν ανθρωπιστικό Διάδομο για την άφηξη των προσφύγων. Αλλιώ τα χέρια σα θα συνεχίσουν να είναι ε, λεκιασμένα με αίμα. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάουταλα για τους πράσινους λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, η Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διασκήψη Κορυφή, η πρώτη που έχει γίνει θα είναι ίσω μια ευκαιρία για να ξανατονίσουμε τη σημασία που έχει το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και μπορεί να βοηθήσει και την συμμόρφωση με το δίκαιο αυτό. Κοιτάξτε όμως τι γίνεται. Είχαμε ήδη αμφιβολίες για το επίπεδο φιλοδοξιών αυτής της διάσκεψης κορφής και ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει ό,τι μπορεί για να μην υποβαθμιστεί αυτό το επίπεδο φιλοδοξίας. Καλό είναι να έχουμε όλους τους εμπλεκόμενους γύρω από ένα τραπέζι αλλά κυρίως το απαραίτητο είναι να υπάρξουν δεσμεύσεις για την βελτίωση της κατάστασης. Οι γιατροί χωρίς σύνορα κρούν τον κόδωνα του κινδύνου γιατί έχουν ήδη αναφέρει ότι θα φύγουν από τη διάσκεψη κορυφής γιατί δεν θα ενισχύσει τις δυσμεύσεις των κρατών μελών να διατηρήσουν <clears throat> το ανθρωπιστικό και προσφυγικό δίκαιο. 75 από τα νοσοκομεία τα οποία υποστηρίζουν έχουν, οι γιατροί σύνορα έχουν βομβαρδιστεί το τελευταίο χρόνο. Αυτό είναι ήδη σκανδαλώδες. Αυξάνεται ο αριθμός των σχολείων και των νοσοκομείων που έτυχαν επιθέσεως. Αυτό είναι όλο και μεγαλύτερη περιφρόνηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Η στόχευση πολιτών και πολιτικών υποδομών είναι έγκλημα πολέμου. Είναι απαραίτητο λοιπόν να εξασφαλίσουμε και την ανεξαρτησία της ανθρωπιστικής βοήθειας και τη σωστή ανακουφιστική βοήθεια. Όλα αυτά τα θέματα πρέπει να αντιμετωπιστούν στη διάσκεψη κορυφή. Πρέπει να βοηθήσουμε και την κατάσταση των γυναικών, των κορισιών και των άλλων ευάλωτων ομάδων που έχουν να αντιμετωπίσουν ανθρωπιστικέ κρίσει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λούντκρεν από την ομάδα EFDD. Ευχαριστώ πολύ. Για πρώτη φορά στην ιστορία πρόκειται να γίνει παγκόσμια ανθρωπιστική διάσκεψη κορυφής. Είναι καλή ιδέα, αλλά διεξάγεται στην Τουρκία. Αυτό θέλει να δείξει ότι υπάρχουν στενές σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία δεν τηρεί τη δημοκρατία, δεν στηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν στηρίζει την ελευθερία έκφρασης, δεν εμφανίζεται δεν είναι καν στην Ευρώπη, είναι στην Ασία και ε, η Τουρκία αναγκάζει την Άγγελα Μέρκελ να ασκήσει δίωξη κατά ενός κομικού και κάνει επιθέσεις σε δημοσιογράφους, σε έναν δημοσιογράφο που ήθελε να επιστρέψει μετά τις διακοπές. Και ισχυρίστηκαν ότι ε, πριν από μερικά χρόνια είχε κάνει ένα tweet που επέκρινε τον κύριο Ερντογάν. Τίποτα δεν είναι ελεύθερο στην Τουρκία. Ε, λοιπόν, αυτοί δεν τηρούν τις αξίες μας καθόλου. Ο κύριος Μπονάνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να ρωτήσω τον Επίτροπο που είναι εδώ παρόν και τον οποίο ευχαριστώ γι' αυτό, πόσο κοστίζει αυτή η διάσκεψη κορυφής για να βοηθήσουμε τις φτωχές χώρες. Γιατί κάθε φορά που μιλάμε, κανείς δεν μας λέει ότι από τα 100 το 80 από αυτά που δίνουμε πηγαίνει για δαπάνες ε, εκπροσώπησης, για να πληρώσουμε τους γραφειοκράτες, για να φτιάξουμε το πλαίσιο, για να βοηθήσουμε τους ε, ε, ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη, μένει πολύ λίγο. Πόσο στοιχίζω επίτροπε, το ξαναρωτώ, αυτή η σάμιτ από όπου, όπου θα φτάσουν οι πάντες. Θα φτάσει και πού πάνε όλοι αυτοί, στην Τουρκία. Είναι σαν, ξέρουμε πόσο δημοκρατική είναι η Τουρκία με τον Ερδογάν, ε, θα ήταν ίσως κόπιμο να φύγουμε γιατί είναι ένας ξεκάθαρος δικτάτορας. Θα, ένα, θα μπορούσε να είναι ο Χίτλερ ε, της επόμενης δεκαετίας. Η Τουρκία είναι σαν να πηγαίνει στο να παίρνει στο τοξικομανής και για να τη βελτιώσει την κατάστασή τους να πάρουμε τον Πάμπλο Εσκομπάρ ως επόπτη τους. Ξέρετε τον Εσκομπάρ που ήταν ένας ε, ένα αφεντικό των ναρκωτικών. Δηλαδή πάμε να κάνουμε συνόδου κορυφή στην Τουρκία. Και εσείς τι κάνετε. Κουβεντιάζετε σε εισαγωγικά ε, για τα ναρκωτικά και φωνάζετε τον Εσκομπάρ να σας βοηθήσει. Μπράβο, μπράβο. Πολύ καλή δουλειά κάνετε. Εξηγήστε στον κόσμο που είναι εδώ πού πετάτε όλα αυτά τα λεφτά. Δεν τα δίνετε στον κόσμο. Τα τρώτε εσεί. Κύριε για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, ακούσαμε ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα και διαφορετική ε, φιλοδοξία και διαφορετικέ απόψει για την διάσκεψη αυτή τη κορυφή. Αν υπάρχει όμω μια συνένεση για το οτιδήποτε, είναι το γεγονός ότι στον κόσμο σήμερα η ανθρωπιστική βοήθεια έχει ξεπεραστεί από την υπερβολική πίεση. Έχουμε έλλειψη κονδυλίων για να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε όλες τις ανθρωπιστικές ανάγκες. Όπως είπε ο κύριος Γκερέρο, είναι εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που χρειάζονται κάποια μορφή ανθρωπιστικής βοήθειας. Έχουμε περισσότερους πρόσφυγες σήμερα από ό,τι μετά από τον Δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο. Δυστυχώς βλέπουμε συγχρόνως να υπάρξει μια μεγάλη αύξηση σε μακροχρόνιες ανθρωπιστικές κρίσεις, μακροχρόνιες μορφές εκτοπισμού που ξεπερνούν τα 25 χρόνια και που ξεπερνούν τα 20 χρόνια στους εσωτερικά εκτοπισμένους. Αλλά λάβουμε τώρα όλα αυτά υπόψη μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε την ανάγκη της παροχής παιδείας εκπαίδευσης, κάτι το οποίο τονίζει και ο Επιτροπός μας. Για αυτές τις μακροχρόνιες κρίσεις τα ανθρωπιστικά συστήματα αυτά από μόνα τους δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων γιατί η μετακίνηση, ο εκτοπισμός δεν είναι ένα πρόβλημα ανθρωπιστικό, αλλά και μια πρόκληση σε επίπεδο αναπτυξιακό και πολιτικό. Δύο λεπτά έχω αν δεν κάνω λάθος. Είναι μια πρόκληση λοιπόν και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχουμε το φαινόμενο των παράτυπων μεταναστών που προκαλείται από τις ανθρωπιστικές κρίσεις αλλά θα πρέπει να λάβουμε και την υπόψη και τη διάσταση ασφαλείας εδώ. Θα ήθελα να απαντήσω στο, στην ανακοίνωση της Κομισιόν η οποία έχει σαν στόχο να μειώσει την εξάρτηση από ανθρωπιστική αρρωγή σε αυτές τις καταστάσεις των ανθρώπων που είναι <clears throat> εκτοπισμένοι, βοηθώντας τους να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή και να συμβάλλουν στη ζωή των κοινωνιών που υποδοχής. Ναι, έχετε δίκιο, ήταν πράγματι δύο λεπτά. Κύριε Κώστα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ελπίζω να ξαναβρει η Ευρώπη τον εαυτό της στην Κωνσταντινούπολη, όντας πρωταγωνίστρια της αλληλεγγύης και της ανθρωπιστικής δράσης ενώπιον της κρίσης των προσφύγων, ιδίως για τους πιο ευάλωτους παιδιά, και μωρά. Γι' αυτό στους ε, σοσιαλιστές ξεκινήσαμε την εκστατεία έντουκα για να παράσχουμε πόρους για την πρόσβαση ανηλίκων στο σχολείο σε συνθήκες επίγοντος χαρακτήρα. Με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Στυλιανίδη γιατί ε, χρήσιμο, επένδυσε 32 εκατομμύρια ευρώ για το 2000, ε, επιπλέον για το 2016 και θα έρθει την άλλη εβδομάδα στη Ρώμη για το ξεκίνημα της καμπάνιας στην Ρώμη. Η εκπαίδευση δεν είναι κάτι μεταγενέστερο, είναι βασικό κομμάτι της υποδοχής, της πρόσβασης, της πρόληψης, της βίας. Γι' αυτό και η ανθεκτικότητα των ε, νέων έχει επιπτώσει στη ζωή. Προτείνουμε και ανθρωπιστικά οκούς διαδρόμους, εκπαιδευτικούς διαδρόμους τους, λέμε για την υποδοχή των φοιτητών μαθητών στην Δυτική Ευρώπη. Είναι σημαντικό και άλλες χώρες, Γερμανία, ε, Ισπανία ίσως να δεχθούν ε, στα μαθήματά τους φοιτητές πρόσφυγες. Ευχαριστώ. Ο κ. Γκέρικε, ένα λεπτό. Σε λίγες μέρες ξεκινάει η παγκόσμια ανθρωπιστική διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στην Κωνσταντινούπολη και εκεί πρέπει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς θα πρέπει να υπενθυμίσουμε και στην Τουρκία τι σημαίνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ανθρωπιστική προσέγγιση. Αυτό το οποίο δεν μπορούμε να δεχτούμε είναι να μην σχολιάζουμε αυτά τα οποία λέει ο Ερντογάν στο πλαίσιο αυτή τη διάσκεψη, όταν υπάρχουν υποχωρήσει σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, κάτι το οποίο το τονίζει και η τελευταία έκθεση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει όλο και περισσότερη περιστολή των ελευθεριών, τη ελευθερία έκφραση και του τύπου. Είναι μεγάλη και η ευθύνη που έχει η Τουρκία για το ρεύμα προσφύγων που πέρασε στην Ελλάδα. Θα πρέπει εμεί ω Ευρωπαίοι να υπενθυμίσουμε ότι οι καλύτεροι στόχοι δεν μπορούν να πετύχουν τίποτα αν δεν υπάρχουν και τα κατάλληλα εργαλεία. Και εκεί θα πρέπει να εστιάσει αυτή η διάσκεψη και έτσι θα μετρηθεί η αξία της, να αντιμετωπίσουν την πείνα της σειράξης και να επενδύσουν στην ε, συγκεκριμένη εφαρμογή των ανθρωπιστικών αξιών. Μία ε, διάσκεψη λοιπόν που να αφορά την πρακτική ανθρωπιστική βοήθεια. Ένα λεπτό κύριε Μπετσέρα Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι επιθέσει ε, σε δομέ και οργανώσει ανθρωπιστική βοήθεια πολλαπλασιάστηκαν τα τελευταία χρόνια. Οι γιατροί χωρί σύνορα μόνο το 2015 κατήγγειλαν 75 επιθέσει σε εγκαταστάσει. Την περασμένη εβδομάδα στο στρατόπεδο προσφύγων στο Σαρμάντα στη Συρία 30 άτομα σκοτώθηκαν σε μια επίθεση που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ω ατύχημα υπάρχει μια επιδείνωση τη συμπεριφορά σου. Ο Υπουργό Εξωτερικών τη Γαλλία σωστά είπε ότι μιλάμε για έγκλημα πολέμου, για έγκλημα κατά τη ανθρωπότητα. Η Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφή ε, για την Ανθρωπιστική σύνοδο πρέπει να χτυπήσει την ατιμορρησία σε διεθνέ επίπεδο και η προστασία των ε, εργαζόμενων τη ανθρωπιστικέ οργανώσει πρέπει να είναι στο κέντρο των δράσεών μα η ασφάλεια και η επιβίωση αυτών που πλήττονται κυρίω θα εξαρτηθεί από αυτή την προϋπόθεση. Ως Ένωση έχουμε την ευθύνη να αυξήσουμε τον ρόλο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου χρησιμοποιώντας τη δυνατότητά μας για να τεθεί τέλος αυτή την απαράδεκτη και εφρικτή κατάσταση. Ευχαριστώ. Ε, είστε ο μιλητής κύριε Φουντσουλίτσα, αλλά είστε και ταυτόχρονα ο Θέλετε να κρατήσετε την μπλε κάρτα. Ε, δεν τηρώ απόλυτα τους κανόνες. Ο κύριος Κοράου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Στην ψηφοφορία της έκθεσης για το World Humanitarian Summit αναγνωρίσαμε ότι η διάσκεψη αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για να μπορέσει η Ευρώπη να αποκτήσει εκ νέου την θέση του πρωταγωνιστή στον τομέα της ανθρωπιστικής αντιμετώπισης. Οι ευχές βέβαια σε τέτοιες διάσκεψεις κορυφής είναι να υπάρξει από κοινού δράση με άλλες έντιμες κυβερνήσεις ούτως ώστε να μπορέσουμε να αποφεύγουμε εφ' εξής δραστηριότητες που οδηγούν σε ανθρωπιστική κρίση. Πρέπει να αναγνωρίσουμε το 80% των κρίσεων προκύπτουν από τις συγκρούσεις αυτών που θέλουν να λύσουν τα προβλήματα ή έτσι λένε. Ε, χώρες ε, μετέχουν εκεί όπως η Σαουδική Αραβία που έχει ε, με τη βοήθεια των, των πωλήσεων όπλων από την Ευρώπη την βασική ευθύνη της ανθρωπιστικής κρίσης στην Ιεμένη. Το ίδιο συμβαίνει και αλλού. Υπάρχει η εγκληματική προσέγγιση της διπλής ή τριπλής επίθεσης. Στον κύριο Στυλιανίδη θέλω να του ζητήσω να δεσμευθεί ότι η Ένωση θα έχει μια σαφή στάση αντίθετα σε μετέχοντες στην διάσκεψη όπως η οδική Αραβία. Ένα λεπτό, ο κύριος Βέντα. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας μας λένε ότι 250 εκατομμύρια άνθρωποι ε, έχουν σχέση με, ε, ε, πλήττονται από μια ανθρωπιστική κρίση. Αυτό οφείλεται σε συγκρούσεις και σε φυσικές και άλλες καταστροφές. Η διάσκεψη κορυφής της Κωνσταντινούπολης θέλει να επισημάνει αυτό το γεγονός και να προσφέρει περισσότερο βοήθεια. Είναι σημαντικό στόχος του ΟΗΕ η οργάνωση μια σειρά ανθρωπιστικών διαβουλεύσεων στην περιοχή. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να είναι το τελευταίο μέσον που πρέπει να χρησιμοποιηθεί όταν όταν τα τοπικά μέσα έχουν ξεπεραστεί. Γι' αυτό πρέπει να στηριχθεί και η τοπική προστασία. Η, παρούσα κρίση έχει μακροχρόνιο χαρακτήρα και γι' αυτό είναι κρίσιμο το θέμα του ε, κενού ανάμεσα στην τρέχουσα βοήθεια και την μακροχρόνια ε, ε, αναπτυξιακή βοήθεια. Ελπίζω ότι η διάσκεψη αυτή κορυφής θα επισημάνει και το θέμα των γυναικών, των παιδιών και των ε, ανθρώπων με αναπηρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπήρχε μπλε κάρτα, κύριε Βέντα. Ε, το δέχεστε, τη δέχεστε, κύριε Ρούμπιτς. Θα ευχαριστούσα τον κύριο Βέντα γιατί έθεσε το ουσιαστικό ερώτημα. Πώς μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και το ερώτημα μου είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να εξασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη αυτονομία των οικογενειακών επιχειρήσεων σε αναπτυσσόμενες χώρες. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε λοιπόν σε αυτούς οι οποίοι βοηθούν τον εαυτό τους και να το συμπεριλάβουμε αυτό στην πολιτική ανάπτυξης ώστε να, δίνε να κάνουμε πιο εύκολο για τις οικογένειες να παράγουν αυτά τα οποία χρειάζονται. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Ρούμπιχ για το ερώτημα αυτό γιατί έχουμε συνεργαστεί σε αυτή την έκθεση, όπως γνωρίζετε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι τόσο σημαντικές για την ενίσχυση των αναπτυσσομένων χωρών. Μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν στο να δημιουργήσουν μια πιο στεναρή και ισχυρή κοινωνία. Αν χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τα εργαλεία της ε, αναπτυξιακής βοήθειας, αυτό θα πρέπει να ευνοεί και την συμμετοχή των ε, οικογενειών αυτών και φυσικά πρέπει να πετύχουμε το στόχο του 0,7% του ΑΕΠ όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι μπορούμε εμείς και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμβάλλουμε στο επιτευχθεί αυτό. Η κυρία Βανερτιάνο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έλεγε ο Επίτροπος Τηλιανίδης ότι θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε το πετραδάκι μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χρειάζεται όμως ένα πετραδάκι κύριε Στυλιανίδη, χρειάζεται κάτι πολύ περισσότερο. Χρειάζεται μια πολιτική δέσμευση, χρειάζονται πόροι, λείπουν τα 40% αυτών που χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε ευφυΐα, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη αποφασιστικότητα ως Ευρωπαϊκή Ένωση για την Κωνσταντινούπολη. Είναι μονάχα ένα πρώτο βήμα. Αν θέλουμε να αλλάξουμε κατεύθυνση στην ανθρωπιστική βοήθεια η οποία οδηγεί σε μια ουσιαστικά γίνεται σε μια κατάσταση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιφρόνησης των ε, δικαιωμάτων των ανθρώπων που βρίσκονται σε βοήθεια. Πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι η Κωνσταντινούπολη αυτή η διάσκεψη σημαίνει τη διαφορά μεταξύ ζωή και θανάτου για πάρα πολλού ανθρώπου και σημαίνει και την αξιοπιστία τη Ευρωπαϊκή Ένωση ω εταίρου ανθρωπιστική βοήθεια στον κόσμο. Ξέρω βέβαια ότι δεν εξαρτάται από το δικό σας χέρι, κύριε Επίτροπε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όμως βρέθηκε παραμερισμένο σε αυτήν τη διάσκεψη. Για όλο το Κοινοβούλιο μονάχα ένα άτομο μπορεί να διαπιστευτεί για να συμμετέχει στις συζητήσεις. Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό και θέλω να υπάρχει μια παρέμβαση από τη δική σας πλευρά για να διορθωθεί αυτό. Η κυρία, Η κυρία Τόμασιτς, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κόσμος δεν έχει αντιμετωπίσει παρόμοιο αριθμό εκτοπισμένων από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα είναι καλή η στιγμή που διεξάγεται αυτή η Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής. Και δεν υπάρχει καλύτερος τόπος να διπραγματοποιηθεί αυτή από την Κωνσταντινούπολη, γιατί η Τουρκία είναι στο επίκεντρο των μεταναστευτικών ροών και είναι εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επίλυση της μεταναστευτικής κρίσης. Η Ευρώπη πρέπει να βοηθήσει την αντιμετώπιση των πηγών πηγών αυτών των κρίσεων και να φροντίζει τους πρόσφυγες. Πιστεύω ότι η διάσκεψη κορυφής θα συνεισφέρει. Δεν μπορώ όμως να παραλείψω να πω ότι κάποιοι θεωρούν ότι αυτές οι ανθρωπιστικές κρίσεις προσφέρονται για εκβιασμούς. Θέλω να επαναλάβω τη θέση μου ε, όσον αφορά το καθεστώς βίζα στην Τουρκία. Χωρίς την ε, τήρηση των τεχνικών κριτηρίων θα ήταν εξαιρετικά ανεύθυνο και θα αποτελούσε και απειλή για τους πολίτες μας κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παέτ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε επισκέφθηκα πριν από λίγε εβδομάδε στο Λίβανο όπου συναντήθηκα και με πρόσφυγες από τη Συρία. Κανένας δεν είπε ότι ήθελε να έρθει στην Ευρώπη. Όλοι ήθελαν να επιστρέψουν στα σπίτια του, στη Συρία για να μπορέσουν να περιμένουν στη γειτονική χώρα για ένα διάστημα και να το κάνουν αυτό με ασφάλεια, ε, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε βασικά αγαθά όπως σχολείο για τα παιδιά τους, δυνατότητα για εργασία και πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη. Αυτό άλλες χώρες όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να το στηρίξουν οικονομικά. Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφή πρέπει να δεσμευτεί ότι θα αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια να μείνουν οι πρόσφυγε κοντά στι αιστείε του. Ένα άλλο πρόβλημα είναι οι υποσχέσει που δίνουν διάφορε χώρε για βοήθεια σε περίπτωση κρίσεων, η οποία όμω δεν έχει προσφερθεί. Α δούμε τα χρήματα που δόθηκαν στην Αϊτή και στον Νεπάλ μετά του σεισμού. Επίση, επίσης εδώ έχει σχέση αυτό και με την ε, κρίση των προσφύγων. Έχουν δοθεί προσ... Ε, αλλά πρέπει να τηρηθούν. Αυτή η παγκόσμια ανθρωπιστική διάσκεψη κορυφής πρέπει να έχει αποτελέσματα και να μην μας απογοητεύσει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πρέντα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το 2015, το Σεπτέμβριο, η Κομισιόν είχε θέσει 7 προτεραιότητες για την ανθρωπιστική δράση. Το ερώτημα που τίθεται τώρα εν ώψη της διάσκεψης, ε, της παγκόσμιας ανθρωπιστικής διάσκεψης είναι Μπορούμε να περάσουμε από την έκφραση καλών προθέσεων σε συγκεκριμένα πράγματα. Νομίζω ότι όπως ε, είπε ο Επίτροπος κ. Στυλιανίδης πρέπει να αναλάβουμε δράση με θαραλέο τρόπο. Η αποφάση και να δώσουμε σαφείς αποφάσεις πρώτον στο έλλειμμα χρηματοδότησης της ανθρωπιστικής βοηθείας δεύτερον, και δεύτερον στην αποτελεσματικότητα του θέματος αυτού. Δεύτερη παρατήρηση για τη σχέση μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και πολιτικών λύσεων για την κρίση. Και εδώ διαφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Κοράο. Δεν νομίζω ότι η ανθρωπιστική βοήθεια μπορεί να υποκαταστήσει τις πολιτικές λύσεις της κρίσης. Από την άλλη, πρέπει, δεν χρειάζεται να αρχίσουμε να κατηγορούμε μόνοι μας στην Ευρώπη. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για το ότι είμαστε οι μεγαλύτεροι δωρητές στον κόσμο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λίτς. Ένα λεπτό. Κύριε, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αυτή η διάσκεψη κορυφής για τα ανθρώπινα για την ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να αποτελέσει ένα ορόσημο. Έχουμε αυτή τη στιγμή πάνω από 250 εκατομμύρια ανθρώπων που πλήττονται από ανθρωπιστικέ κρίσει. 60 εκατομμύρια λόγω πολέμων, συγκρούσεων και φυσικών καταστροφών έχουν αναγκαστεί να φύγουν από την ε, Εστία του, Η μισή από αυτού είναι παιδιά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κάτι μέλη θα δείξουν αλληλεγγύη και ευθύνη μονάχα αν δώσουν το καλό παράδειγμα σε αυτή τη διάσκεψη κορυφή με το να τηρήσουν τι υποσχέσει του για χρηματοδότηση. Ένα καλό παράδειγμα για αυτέ τι δυνατότητες είναι η λεγόμενη πρωτοβουλία Εντούκο τη ομάδα μου που λέει ότι αντί για 2% 4% τη ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να πηγαίνει για εκπαίδευση και κατάρτιση θα θέλαμε ο, η Κομισιόν να συμπεριλάβει αυτή την πρόταση στον επόμενο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ω εισηγητή για την ε, ανθρωπιστική βοήθεια στον προπολογισμό 2016, έχω τονίσει ότι πρέπει να δοθούν 26 εκατομμύρια περισσότερο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να κάνουν ό,τι μπορούν ώστε να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία Εντούκα μέσα στην ανθρωπιστική βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Ο Κόμπατσεφ, για ένα λεπτό, έχει το Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Η παγκόσμια διάσκεψη, ανθρωπιστική διάσκεψη κορυφής θα δημιουργήσει ένα βιώσιμο πλαίσιο ανθρωπιστικής βοήθειας. Όπως ακριβώς ε, χρειάζονται πάνω από 110 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο. Ελπίζω ότι αυτή η διάσκεψη θα έχει καλύτερα αποτελέσματα από οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια που έχει γίνει. Ένα από τα θέματα στην ημερήσια διάταξη είναι το θέμα της χρηματοδότησης της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ως εισηγήτρια του... Ε, ως εισηγητής του ε, ΕΛΚ για το θέμα της ε, ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ως μόνιμος εισηγητής για τη, στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θέλω να επιμείνω για τρία, σε τρία πράγματα. Πιο αποτελεσματική προσπάθεια για τη διάλυση των τρομοκρατικών δικτύων. Δεύτερον, να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στο διαπολιτισμικό διάλογο. Τρίτον, η η προσφορά ανθρωπίνων και χρηματικών ε, πόρων για την διατήρηση και την στήριξη αρχών όπως ε, η ένωμη τάξη και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η Τουρκία είναι οικοδεσπότης για τις διάσκεψεις αυτής. Θα πρέπει να προσπαθήσει για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που έχουν ανάγκη σε ολόκληρο τον κόσμο. Δόθηκε η δυνατότητα στην Τουρκία να είναι οικοδεσπότης πριν η Ευρώπη και η Τουρκία πλημμυρίσουν από τις ροές των προσφύγων έχει κάποιο συμβολισμό το γεγονός ότι ο κόσμος θα συναντηθεί στην Κωνσταντινούπολη για να αντιμετωπίσει συγκεκριμένες λύσεις και να ενισχύσει την θέση της Ευρώπης ως βασικό δωρητής. Ευχαριστώ. Επόμενο κ. Φροντσολίκα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, διάσκεψη κορυφής θα κάνει σημαντικά βήματα μπροστά για να εντοπίσει λύσεις για να αναμορφώσει το ανθρωπιστικό σύστημα. Κύριε Επίτροπε, είναι θέμα εν τέλει του πόσο φιλόδοξη είναι η Ένωση. Εμείς ως Ένωση πρέπει να έρθουμε με συγκεκριμένες προτάσεις για, μια, για ένα νέο πραγματικό ανθρωπιστικό σύστημα στον κόσμο. Ούτως ώστε να αναλάβουν όλες οι χώρες Ένωσης πλήρη ευθύνη για το θέμα αυτό και να κάνουν την ανθρωπιστική βοήθεια λιγότερο επικίνδυνη. Για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς είναι αναγκαίο να υπάρχει κοινή συνεννόηση μεταξύ των εμπλεκόμενων, ε, να υπάρξει λογοδοσία, διαφάνεια και να προλαμβάνουμε τους κινδύνους κάνοντας σαφή κοινό προγραμματισμό. Ευχαριστώ. Κύριος Αντάκτουσον, ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, η Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής της Κωνσταντινούπολης λαμβάνει χώρα σε μια πολύ σημαντική στιγμή. Οι συμμετέχοντες θα προσπαθήσουν να βάλουν στην καλύτερη δυνατή χρήση την ανθρωπιστική βοήθεια. 250 εκατομμύρια άτομα έχει υπολογιστεί ότι χρειάζονται ε, ανθρωπιστική βοήθεια σε 37 χώρες. Οι Γιαζίδη και πολλοί άλλοι είναι από τους πιο εκτεθειμένους. Όταν πήγα πρόσφατα στο Ιράκ ε, διαπίστωσα πόσο σημαντική η συνεισφορά, είναι η συνεισφορά της Ευρώπης. Βεβαίως περισσότερα μπορούν και πρέπει να γίνουν. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι η αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνδεθεί πιο στενά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ένα παράδειγμα είναι η στήριξη προς την Ερυθρέα, η οποία παρατάθηκε πέρυσι χωρίς καμία απέτηση για δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Εδώ πρέπει να μάθουμε από, τα, από την εμπειρία μας. Η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα στην ε, ευρωπαϊκή συνεργασία και τα θέματα, στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σίλβα Περέιρα για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, αντιμετωπίζουμε τόσα ανθρώπινα δράματα ανθρωπιστικού χαρακτήρα και όχι μόνο το θέμα, το θέμα των προσφύγων, αλλά 125 εκατομμύρια ατόμων που ζητούν βοήθεια. Αυτό το οποίο θα έπρεπε να υπάρχει από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι μια μεγάλη κινητοποίηση πολιτικής θέλησης και πόρων, ώστε η επόμενη ώστε η επικείμενη διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης να δώσει μια συγκεκριμένη απάντηση από την πλευρά της διεθνούς κοινότητας. Δυστυχώς, οι προπαρασκευαστικές ε, εργασίες σημαίνουν ότι θα είναι πολύ λιγότερα τα αποτελέσματα από αυτά. Χρειάζεται μεγαλύτερη ευθύνη και μεγαλύτερη ηγετική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό θα πρέπει να γίνει μέσα από υποδειγματικές δεσμεύσεις. Κύριε Πίτροπε, γνωρίζουμε τη δική σας προσωπική προσήλωση στα θέματα αυτά, αλλά χρειάζεται ένα πραγματικός οδικός χάρτης για την ανθρωπιστική βοήθεια, το οποίο σημαίνει και μια σημαντική διεύρυνση των κονδυλίων για την ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την αξιοπρέπεια αυτών των ανθρώπων. Ο κύριος Σένφελτ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η ιστορία των ανθρωπιστικών ενεργειών είναι μακρά όπως και η ιστορία της ανθρωπότητας. Έχουν αλλάξει όμως οι συνθήκες και γι' αυτό θα πρέπει να χαιρόμαστε και να εξασφαλίσουμε ότι προσαρμαζόμαστε στην πραγματικότητα. Χρειάζεται λοιπόν μία ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας για τα 120 εκατομμύρια ανθρώπων που οι μισοί από αυτούς έχουν εκτοπιστεί λόγω ένοπλων συγκρούσεων. Η, η ανθρωπότητα χρειάζεται νέες μορφές ανθρωπιστικού δικαίου. Θα πρέπει να μπορέσει να ενημερωθεί το πεπαλεωμένο πεπαλαιωμένο σύστημα που χρησιμοποιούμε μέσα στις δομές των Ηνωμένων Εθνών. Περιμένω ότι αυτή η διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης θα συμβάλλει στο να υπάρξει μια λύση για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και την έλλειψη συντονισμού και την έλλειψη κονδυλίων μεταξύ των φορέων του ΟΗΕ και με τον τρόπο αυτό επίσης να μπορέσει να υπάρξει και μια πραγματική συμμετοχή και χορηγών όχι από τη Δύση μονάχα. Word για ένα λεπτό. Η παγκόσμια διάσκεψη κορυφής έχει στόχο να αλλάξει την προσέγγιση της, του κόσμου στην ανθρωπιστική βοήθεια. Η Ευρώπη θα είναι μπροστά στη συζήτηση αυτή. Από την οπτική της Βρετανίας και εν ώψη και του δημοψηφίσματος πρέπει να επαξετάσουμε τη θέση μας στον κόσμο. Και πιστεύω ότι μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας μπορούμε να αναμορφώσουμε προς τα βέλτιο την παγκόσμια ημερήσια διάταξη. Αν θέλουμε να οδηγήσουμε την παγκόσμια κοινότητα σε έναν κόσμο με περισσότερη συμπόνια, θα πρέπει να ενισχύσουμε ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ταυτόχρονα με την ε, ε, εξουσία πρέπει να έχουμε και τις ευθύνες μας πρέπει να τηρούμε τις αρχές μας σε όλες τις πολιτικές προς τα έξω ακόμα και υποπίεση η ανθρωπιστική βοήθεια στα θύματα της ανθρωπιστικής κρίσης σημαίνει ότι δεν μπορεί να τα βρίσκουμε με τα καθεστώτα που διαπράττουν αυτά τα, τα εγκλήματα όλα, ε, ε, η διαδικασία του χαρτούμ για παράδειγμα πρέπει να εφαρμόζεται παντού σε όλους τους ε, ε κανονισμούς, σε όλους τις προσεγγίσεις. Ο κύριος Μπόκοβιτς στη διαδικασία Catch the Eye. Ευχαριστώ πολύ. Φυσικά η Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορφής έρχεται πραγματοποιεί την κατάλληλη στιγμή. Γιατί, όπως ακούσαμε, ποτέ δεν υπήρχαν τόσο πολλοί που να χρειάζονται τη βοήθειά μας. Ποτέ δεν υπήρχαν τόσο εκτοπισμένοι στον κόσμο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η λύση που επιδιώκουμε έχει σχέση με αυτό που είπε η Υπουργό στην εισαγωγική της ομιλία. Πρέπει να εντοπίσουμε τις αιτίε των συγκρούσεων, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αντικειμενικά μια πολιτική ανθρώπινη πρέπει οι συγκρούσεις να λύνονται ειρηνικά και όχι με περαιτέρω διαίρεση του κόσμου. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δείξει στον κόσμο τις αξίες της, να επιτρέψουμε στον κόσμο να ζει με αξιοπρέπεια. Πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους στην Αφρική, την Ασία, τη Μέση Ανατολή. Και αυτό θα βοηθήσει και την ίδια την Ευρώπη. Γιατί πού θα πάνε οι ε, ε, πρόσφυγες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας που, είναι, που θα είναι παρούσα στην ε, Κωνσταντινούπολη. Αυτό είναι ηρωνικό ότι γίνεται στην Τουρκία. Αλλά δεν έχουμε καταφέρει παρόλα αυτά να αντιμετωπίσουμε τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά από τον πόλεμο και την τρομοκρατία στο Ιράκ, στη Συρία και τη Λιβύη και που είναι και και του ρεύμα που προέρχεται από την αθλειότητα άλλων χωρών της ε, Αφρικής. Η Τουρκία παραβιάζει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για, την, ε, για τους πρόσφυγες και παραβιάζει και τις θεμελιώδεις αρχές του ανθρωπιστικού δικαίου. Είναι ντροπή για την Ευρώπη που και η ίδια η Ευρώπη παραβιάζει στα hot spots της Ελλάδος έχει τους ε, σορευμένους ε, πρόσφυγες ακόμα και γυναίκες και παιδιά ανήλικα. Όλα αυτά που γίνονται είναι απαράδεκτα. Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι και πάλι μια άσκηση υποκρισίας εάν συνεχίσουμε τις πολιτικές λιτότητος που όλη την περιοχή της Μεσογείου. Και εξακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίζει τις προσπάθειες να δεν κάνει καμιά προσπάθεια να ξεπεράσει τις δικτατορικές κυβερνήσεις της περιοχής. Ευχαριστώ, λέγει πρόεδρος. Ο κύριος Μαριάς. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι οξύμορο η πρώτη παγκόσμια ανθρωπιστική διάσκεψη κορυφή να λαμβάνει χώρα στην Κωνσταντινούπολη. Μια πόλη στην οποία οι διαδηλώσει τη 1 η Μαΐου πνίγηκαν στο αίμα. Είναι οξύμορο το μεγαλύτερο γεγονό στη φετινή ατζέντα του ΟΗΕ να φιλοξενείται σε ένα κράτο στην Τουρκία, που παραβιάζει κατάδειλα τα κοινωνικά δικαιώματα, τροφοδοτεί αιματηρού πολέμου, καταπιέζει μειονότητε και πολιτικέ πεπιθήσει στα πλαίσια της διάσκεψης η ευρωπαϊκή ένωση οφείλει να δώσει απτές απαντήσεις στην μείζωνα ανθρωπιστική κρίση που βιώνει σήμερα ο λαός της συρίας με ευθύνη της τουρκίας μια ανθρωπιστική κρίση που μεταφέρεται στην ευρώπη και ιδιαίτερα στην ελλάδα και θα συνεχίσει να υπάρχει όσο η ευρωπαϊκή ένωση θα ανέχεται και θα αφήνει τον ΤΑΕΣ και τους υποστηρικτές του να συνεχίζουν το εγκληματικό τους έργο η ανθρωπιστική κρίση όμως δεν πλήττει μόνο τους πρόσφυγες πλήττει και τον ελληνικό λαό που έχοντας φτωχοποιηθεί από τα μνημόνια και την τρόικα δεν μπορεί πλέον να φιλοξενήσει άλλους πρόσφυγες. πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια διεθνή απάντηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και πρόβλημα και οι πλούσιες χώρε, όχι μόνο στην ευρώπη να συνδράμουν αποφασιστικά στην αντιμετώπιση του. ευχαριστώ. Ε, Κύριε Σόγκορ, ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι γεγονός ότι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν θυγεί από φυσικές καταστροφές αλλά κυρίως από βίες ένοπλες συγκρούσεις έχει αυξήσει. Ποτέ δεν είχαμε τόσου πολλού ανθρώπου που έχουν εκτοπιστεί από τι αιστείε του μετά το δεύτερο παγκοσμίο πόλεμο. Αυτό δικαιολογεί την οργάνωση μια παγκόσμια ανθρωπιστική διάσκεψη. Αλλά αν λάβουμε υπόψη το πόσοι άνθρωποι χρειάζονται αυτή τη βοήθεια και δεν τη λαμβάνουν, βλέπουμε αυτούς, βλέπουμε το κόσμο να είναι διχασμένο σε δύο κομμάτια. Αυτούς οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν, αλλά δεν το κάνουν και άλλους οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα. Δεν είναι επαρκή οι βοήθειες που δίνονται από του χορηγού, Χρειαζόμαστε παγκόσμια συνεργασία για τα θέματα αυτά Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ανακουφίσουμε τα βάσανα αυτών των ανθρώπων που προσπαθούν να ξεφύγουν από την τρομοκρατία και τις βίαιες συγκρούσεις. Υπάρχει και η <clears throat> ταχεία δημογραφική ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες περιοχές που είναι ένα πρόσθετο πρόβλημα. Κύριε Τιέγγε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα βλέπουμε τη μεγαλύτερη μετακίνηση ανδρών, γυναικών και παιδιών μετά το Δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο. 250 εκατομμύρια άτομα κινούνται, 60 εκατομμύρια πρόσφυγες ανά τον κόσμο. Έχουμε μπροστά μας μια πραγματική ανθρωπιστική κρίση σε πλανητικό επίπεδο. Ο κόσμος φεύγει τον πόλεμο, τη φτώχεια, την αλλαγή του κλίματος. Ευπρόσδεκτη λοιπόν η διάσκεψη κορυφής, διότι μπορεί να βάλουμε κάποια σημαντικά θέματα στο κέντρο των συζητήσεων. Την επανεξέταση, για παράδειγμα, της χρήσης της ανθρωπιστικής βοήθειας, προς, πηγαίνοντας προς πολιτικές ανάπτυξης που θα πρέπει να προσβλέπουν μέσω και μακροπρόθεσμα τις ε, αιτίες, τις πραγματικές αιτίες που οδηγούν στη μετακίνηση των ανθρώπων. Πολιτικές πρόληψης, που πρέπει να αντιμετωπίζουν και επίγοντα, επίγοντα περιστατικά όπως τον ανθρωπιστικό διάδρομο, την αντιμετώπιση καταστάσεων που όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και εκτός, στο Λίβανο, στη Συρία. Πρέπει να προχωρήσουμε σε μια πολιτική πρόληψη αποφεύγοντας την πολιτική αντιμετώπιση κρίσεων και μόνο. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται η διαδικασία Catch the Ο κύριος Τηλιανίδης έχει το λόγο τώρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πολύ επικοδομητική και παραγωγική συζήτηση. Πάντοτε εκτιμώ τις θέσεις ε, και τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίως καθώς προετοιμαζόμαστε για τη μοναδική αυτή πολυμερή εκδήλωση, την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής. Και γι' αυτό επέμενα στο να αυξηθούν οι θέσεις για το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου στην διάσκεψη. Καταβάλαμε ό, μεγάλη προσπάθεια ώστε να εκπροσωπηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκεί και σήμερα μπορούμε να πούμε με χαρά ότι έχουμε εξασφαλίσει δύο επιπλέον θέσεις στην αντιπροσωπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι προτεραιότητες μας είναι κοινέ. Περισσότερη αποτελεσματικότητα, περισσότερη αποδοτικότητα του ανθρωπιστικού συστήματος, ένα σεβασμό για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και βεβαίως και για τις ανθρωπιστικές ε, αρχές. Περισσότερη υποστήριξη για τις καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Για το λόγο αυτό υπάρχει στενή αυτή η συνεργασία. Επειδή είμαστε δίπλα-δίπλα. Η διάσκεψη αυτή κορυφής θα ολοκληρώσει έναν κύκλο διάσκεψη για τους στόχους της ε, χιλιετίας ε, η, της Αντίσα Μπέμπα, η COP21 έχουν προσφέρει ένα όραμα για το μέλλον. Τα αποτελέσματά τους αποτελούν ένα ισχυρό πλαίσιο για να προχωρήσουμε στο μέλλον. Όμως η πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν πλέον στραφούμε προς τις, τους φτωχότερους και τους πλέον ευάλωτους για να τους βοηθήσουμε να ζήσουν καλύτερα. Αυτό είναι, αυτός είναι ο σκοπός της Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης Κορυφής. Το 2030 ελπίζω ότι κοιτώντας πίσω θα μπορέσουμε να πούμε ότι λόγω αυτής της διάσκεψης άλλαξε η κατάσταση. Η, η μακρά περίοδος διαβουλεύσεων επέτρεψε σε όλους να εκφραστούν από τους ηγέτες μέχρι τα μέλη των πληττόμενων κοινοτήτων ε, τους ακαδημαϊκούς, τον ιδιωτικό τομέα. Συμμετείχαν χιλιάδες από ολόκληρο τον κόσμο και ε, δημιουργήθηκε ένας νέος τρόπος προώθησης των πιο δύσκολων καταστάσεων και δημιουργήθηκε μία όθηση η οποία ελπίζουμε ότι θα οδηγήσει σε συστημικές αλλαγές για τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκρινόμαστε και θα ανακάμπτουμε αποκρίσεις. Ελπίζω ότι μέχρι το 2030 θα χρειάζεται να προσφέρουμε λιγότερη ε, βοήθεια για αυτούς, σε ανθρώπους που χρειάζεται για να σώσουμε τη ζωή ανθρώπων. Στην διάσκεψη κορφής θα εγκριθεί μια δεύτερη ομάδα συμπερασμάτων με την Προεδρία. Έχουμε συνεργαστεί θα μας καθοδηγήσει για να αναλάβουμε δεσμεύσεις και στη διάσκεψη αλλά και πέρα από αυτήν. Όπως πάντα υπολογίζω στη συνεχή στήριξη και συνεργασία σας κατά την συνέχιση αυτής της προσπάθειας έτσι ώστε να έχουμε ηγετική θέση και να μπορέσουμε να ε, τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία από το Συμβούλιο θα κλείσει τη σχετική συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η παγκόσμια διάσκεψη κορυφή είναι μια αφετηρία του από την ούτως ώστε η παγκόσμια κοινότητα να αποκαταστήσει την, τον ανθρωπισμό, όπως είπε ο γενικό Γραμματέα του ΙΕ πολλέ φορές. Ελπίζουμε να υπάρχουν ουσιαστικές και πολλές δεσμεύσεις στο ανώτερο δυνατό επίπεδο από όλους τους εμπλεκόμενους ε, παράγοντες και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα αντιμετωπιστεί η διάσκεψη ως ένα, μια εκδήλωση όπου κυριαρχούν οι δυτικέ θέσεις. Γι' αυτό υπάρχει και συντονισμός από πολλά κράτη εκτός Ένωσης, ιδίως εκτός Ένωσης θα έλεγα. Και συμφωνώ μαζί σας ότι από την πρώτη μέρα μετά την διάσκεψη κορυφής θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε σοβαροί σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε. Ως Προεδρία του Συμβουλίου εμείς ε, παίζουμε, διαδραματίζουμε το ρόλο που μας στο πλαίσιο αυτό και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και τις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και την Επιτροπή. Σας ευχαριστώ τα Η συζήτηση έχει κλείσει και το θέμα αυτό